Bonjour. Καλησπέρα σα. Ε, μία ανακοίνωση από του διερμηνεί. Οι διερμηνεί σα ενημερώνουν ότι συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα κινητοποίηση μα για τι συνθήκε εργασία, γιατί η δίκηση δεν έχει έρθει σε καμία επαφή μαζί μα για την επίλυση τη εργασιακή διένεξη. Σα ενημερώνουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν θα επηρεαστεί από τι εν λόγω κινητοποίησει. Λοιπόν, περνάμε στην ημερησία διάταξη. Συνθήκε εργασία σε τομεί παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εκμετάλλευση. Ε, και έχουμε προσκεκλημένο τον ε, κύριο Ρέμκο ε, Μπρόκερ, καθηγητή, ο οποίος ε, είναι καθηγητής κορεατικών σπουδών στο Λάιντεν, στις κατοχώρες. την κυρία Οτέγγι που είναι υπεύθυνη κατάρτισης του Ισπανικού Συνδικάτου Κομισιόνε Σομπρέρας, τον κύριο Ντερίνκ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έρευνα ε, στον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βιέννη και τον κύριο Τζουζέπε Ιουλιάνο, μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχουμε διαθέσιμες όλες τις γλώσσες, εκτός από τα βουλγαρικά, τα μαλτεζικά και τα κροατικά. Ο κάθε ομιλητής ε, μπορεί να μιλήσει για 10 λεπτά περίπου. Και στη συνέχεια θα έχουμε ερωταπαντήσεις από τους βουλευτές. Και να δούμε αν θα υπάρξουν ερωτήσεις και βουλευτές. Λοιπόν, να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπρούκερ. Oui. Sì, buonasera a tutti. Sono una Κύριε Μπρούκερ, είναι μια δημόσια ακρόαση όπου θα έπρεπε να συμμετέχουν ε, οι συνάδελφοι ευρωβουλευτέ, λέει η κυρία Ατζέα. Εγώ ζητώ συγγνώμη εξ ονόματο ε, όλων γιατί λυπάμαι και τρέπομαι που είμαι εδώ μόνη μου. Δεν ξέρω αν ε, είναι αυτή μια συμπεριφορά που να δείχνει σεβασμό απέναντι σε προσκεκλημένους που έρχονται να μας μιλήσουν για ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να, για το οποίο θα πρέπει να αναλυφθεί δράση για την επίλυσή του. Εμένα με ενδιαφέρει να αντιμετωπίζω θέματα όπως έχουν να κάνουν με την καταργαστική εργασία που ενδιαφέρουν και τα 28 κράτη-μέλη και αφορούν εκατομμύρια άτομα. Και αν σκεφτούμε την περίπτωση της Ιταλίας, ε, οι άνθρωποι αυτοί ζουν ε, υπό καθεστώς και μάλιστα πολλές φορές χάνουν και τη ζωή τους ε, λόγω των συνθηκών εργασίας τους, ε, χωρίς δικαιώματα, χωρίς καμία προστασία, με μια εκμετάλλευση ε, που πάει πολύ πιο πέρα από τα δεινά. Και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος όλων όσων απουσιάζουν. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας και ως έκτακτος πρόεδρος και εγώ θέλω να σας ε, ζητήσω συγγνώμη. Δυστυχώς δεν είχε προβλεφθεί και εγώ στις 3.30 θα πρέπει να πάω σε μια επιτροπή όπου είμαι συντονιστής για θέματα τρομοκρατίας. Και υπάρχει φυσικά αυτός ο κίνδυνος της εκμετάλλευσης στην Ιταλία, ε, παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα δώσω λοιπόν ε, κατευθείαν το λόγο στον καθηγητή Μπρόκερ. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ να μιλήσω για αυτά τα εξωτικά ζητήματα εκμετάλλευση ε, των ε, εργαζομένων από την Κορέα ή από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα ε, με το οποίο ασχοληθήκαμε εμείς τα τρία τελευταία χρόνια. Και θα αναφερθώ, τρία, θα αναφερθώ σε τρία σημαντικά σημεία για αυτή τη συνεδρίαση. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι φαίνεται να είναι νόμιμοι είναι νόμιμα παρόντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σημαίνει ότι έχουν άδειε εργασία και θεωρήσει εργασία. και φυσικά αυτό θα έπρεπε να συμβάλλει στην καταπολέμηση εκμετάλλευση, όμως στην πράξη δεν συμβαίνει. Και ε, βλέπετε ε, ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κυρίως στην Πολωνία επικέντρωσαμε την ευρά μας, αλλά δεν πρόκειται μόνο για την Πολωνία και προσαρμόζονται σε συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη έχουμε υπεργολαβία, εργαζομένους ε, στον κατασκευαστικό τομέα και υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι που είναι σε παράνομη κατάσταση, σε μη παράνομη κατάσταση, αλλά και σε νόμιμη κατάσταση. Δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να καθορίσουμε το συνολικό αριθμό των εργαζομένων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα στατιστικά στοιχεία που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη. Αλλά στην πράξη, τέλο πάντων, δεν μπόρεσαν να μας τα δώσουν. Το γεγονός ότι είναι νόμιμοι αυτοί οι εργαζόμενοι και έχουν θεωρήσεις και άδειες εργασίας ε, καθιστά πολύπλοκο το θέμα, την εικόνα, γιατί ε, όχι μόνο γιατί ε, βρίσκουν δουλειά και κατασκευές αλλά έχουμε και υπεργολαβία, αλλά τους ε, βρίσκουμε και να εργάζονται σε κάποιες εταιρείες με τοπική έδρα και μάλιστα οι εταιρείε αυτές λαμβάνουν ακόμη και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους από τη Βόρεια Κορέα. Και από ό,τι φαίνεται, είναι μια συμφωνία μεταξύ των ε, κρατών μελών και της ε, Λαϊκής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας. Και έρχομαι σε δεύτερο, στο δεύτερο σημείο ότι ε, τι συμβαίνει σε αυτούς, ε, ό,τι συμβαίνει σε αυτούς είναι παράνομο γιατί ξέρουμε ε, η Βόρεια Κορέα είναι ένα αυταρχικό δεκτατορικό κράτος και οι εργαζόμενοι που στέλνει εδώ δεν έχουν λόγο για το τι τους συμβαίνει, δεν ξέρουν καν σε ποια χώρα θα τους στείλουν, τους παίρνουν το διαβατήριο, δεν έχουν τίποτα σύμβαση εργασία, δεν έχουν ε, λογαριασμό στην τράπεζα και φυσικά δεν μπορούν ε, να πούν τίποτα σε σχέση με την κατάστασή Του Μπορεί να χρειάζεται να εργάζονται 12-16 ώρες τη μέρα και το κάνουν και φυσικά δεν μπορούν να διαβάσουν εφημερίδε, ε, ούτε να έχουν προσθέσει στο διαδίκτυο, ούτε να μιλήσουν στου ντόπιου και δεν έχουν επιλογή παρά να υπακούσουν. Και στην πράξη θα βρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνται σε ομάδε, ε, είναι μόνο μεταξύ του, είναι πολύ καλοί εργαζόμενοι, γιατί δεν λένε ποτέ όχι, δεν φέρνουν καμία αντίρρηση στο ότι του ζητάνε, δεν έχουν τραπεζικού λογαριασμού και αν πληρώνονται, πληρώνονται ίσα ίσα για να αγοράσουν τσιγάρα και μπύρε. και φυσικά τους αφαιρούν διαφορά έξοδα από το μισθό τους. Μένουν 3-5 έτη, μερικές φορές και περισσότερο. Οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες ε, στο βαθμό που ε, σκοτώνονται άνθρωποι. Από το 2014 είχαμε διάφορα μέτρα γιατί το κράτος της που είναι υπεύθυνο για τους ανθρώπους αυτούς ε, δεν ήθελε να επενδύσει σε θέματα ασφαλείας και μετά το 2014 αυτό άλλαξε, όμως και πάλι είναι δύσκολη κατάσταση και έχουν τις πιο δύσκολες και επικίνδυνε δουλειές. Πολύ συχνά έχουμε τυχήματα δηλαδή. Και υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα που σχετίζεται με αυτό, κάτι που είναι παράνομο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η εξαγωγή ε, του ε, ιδεολογικού συστήματος της καταστολής και καταπίεσης της Βόρειας Κορέας. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε 50-80 άτομα που δουλεύουν σε ένα μέρος και αναγκάζονται να υπακούσουν στους ίδιους κανόνες που θα ίσχυαν στη Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, θα ε, πρέπει να ασκούν αυτοκριτική, θα πρέπει να ομολογούν πίστη στο καθεστώς και φυσικά αυτό διατηρεί την ομάδα ενωμένη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ όχι αδύνατο για αυτούς, ε, να αντισταθούν ε, στην εκμετάλλευση στην οποία είναι εκτιθυμένοι. Γιατί γενικά τι είδαμε ότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουν 12-16 ώρες τη μέρα και μερικές φορές και 24 ώρες συνεχόμενες. Πριν το χάρη στα ναυπηγεία στον κατασκευαστικό τομέα. Πρόκειται για επικίνδυνη δουλειά και φυσικά αν κουραστεί κάποιος μπορεί να γίνουν κατηχήματα. Όμως ε, δεν μπορείς να πεις όχι στο λόγω του συστήματος όπως σε συνοδεύει και ε, στέλνονται άνθρωποι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ένας τόπος που θέλουν ε, να έρθουν ε, πολλοί άνθρωποι και πολλές φορές αφήνουν πίσω την οικογένειά τους, ε, τη γυναίκα τους και δύο παιδιά συνήθως και ουσιαστικά είναι σαν όμοιροι. Αν ε, επιλέξουν ε, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως υπήκοοι τρίτης χώρας, υπάλληλοι τρίτης χώρας, οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να μπουν σε κάποιο συνδικάτο, να δημιουργήσουν συνδικάτο ή να παρατηθούν, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν, η οικογένεια υποφέρει. Φτάνω στο τρίτο σημείο, το τελευταίο σημείο. Έχουμε μέτρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουμε την εργασιακή εκμετάλλευση και όπως ανέφερα στο πρώτο μου σημείο, καθώς αυτή η η τρίτης χώρας ε, είναι εδώ με νόμιμες ε, θεωρήσεις και άδειες ε, εργασίας, δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να κάνουμε κάτι. Στην πράξη όμως δεν φαίνεται να ισχύει αυτό. Βλέπουμε διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο είναι το σενάριο στο οποίο η επιθεώρηση εργασίας κάνει τη δουλειά της σωστά, κάνει τις επιθεωρήσεις ε, και συλλέγει αποδείξεις ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι παραβιάζεται όλη η νομοθεσία. Το πρόβλημα που βρήκαμε στη συνέχεια είναι ότι οι επιθεωρήσει εργασία συχνά δεν έχουν την εξουσία για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έτσι στην πράξη αφού επιβάλλουν ε, πρόστιμα που είναι συμβολικά γιατί συνήθω είναι πολύ χαμηλά, όλα συνεχίζουν όπως και πριν. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Κατόπιν υπάρχει το δεύτερο σενάριο που έχουμε δει, αφού δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση το 2016 και είχαμε έτσι πολύ μεγάλη αντίδραση από τα μέσα μας εξενημέρωσης. Είδαμε ότι ασκήθηκε πολιτική μείωση στους ε, επιθερωτές εργασίας και τι βρήκαμε ότι αφενός οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή συνεχίζεται η εκμετάλλευση, πρέπει να δουλεύουν πολλές ώρες, δεν παίρνουν ε, άδεια, ε, μπορεί να παίρνουν άδεια έξι ώρες σε δύο εβδομάδες, δεν μπορούσαν να πάρουν αναρωτική, γιατί αλλιώς δεν πληρώνονται, δεν μπορούν ε, να παρετηθούν και πληρώνονται περίπου 50 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο και φυσικά δεν μπορούν να, να προβούν σε ανυπακοή. Και ταυτόχρονα βλέπουμε εκθέσει τη επιθεώρηση εργασία που έλεγε ότι όλα ήταν πολύ καλά γιατί μόλις είχαν ε, ελέγξει ε, την, ε, τα χαρτιά, την πραγματικότητα των χαρτιών, ότι είχαμε δηλαδή εντελώς νόμιμες θεωρήσεις και τις εργασίας. Όμως οι επιθεωρητές δεν ε, πήγαν ε, στα ίδια τα μέρη όπου έλαβαν χώρα η εκμετάλλευση, λάμβανε χώρα η εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν δύο πραγματικότητε, ή μάλλον μία διαφορετική πραγματικότητα, η πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών, οι κοτρεί τη χώρα που δεν μπορούν να φύγουν και πρέπει να, πούν, ε, πρέπει να κάνουν ό,τι λένε οι εκμεταλλευτέ του αφενό και αφετέρου έχουμε την πραγματικότητα στα χαρτιά που λέει ότι τίποτα δεν συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν άδειε εργασία και θεωρήσεις. Και μάλιστα υπάρχει και μια ακόμη πιο ανησυχητική προοπτική. Είναι εξή. Ε, εξετάσαμε τις θεωρήσεις και τις άδειες εργασίας που δόθηκαν από το κράτος μέλος και βρήκαμε όμως ότι οι Βορειοκορεάτες ε, έχουν ε, μακροπρόθεσμε άδειε παραμονή ε, και εργασία και δεν εμφανίζονται στι επομένως Επομένω, δεν ξέρουμε πόσοι από αυτού είναι εδώ. Αν έχουν, παραδείγματο χάρη, καθεστώ μακροπρόθεσμη άδεια παραμονή, θα εξαιρεθούν από το καθεστώ επιβολή κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ, γιατί αυτό είναι ένα σενάριο που κανένα δεν είχε προβλέψει. Νομίζω ξανεμίστηκε ο χρόνο μου. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσα να τη μιλήσει και λίγο παραπάνω. Εγώ προτείνω να ακούσουμε τι ερωτήσει από τη Λάουρα. Φαντάζομαι δεν έχει Λάουρα ερωτήσει. Δεν έχει. Μετά λέει. Συνολικά. Εγώ έχω. Είπατε ότι έχουν μια διαργασία σε αυτοί οι άνθρωποι που είναι νόμιμοι. Τρία με πέντε χρόνια λέτε και εργάζονται 12 με 15 ώρες τη μέρα. Έχουμε την τροπολογική της οδηγίας για τους απασπασμένους οι προσωρινά ω εργαζόμενοι μπορούν να έρθουν από τον Ισημερινό, ε, περνάνε στην Ισπανία και μπορούν να έρθουν να δουλέψουν για παράδειγμα στη Γαλλία. Τα έχετε μελετήσει πολύ καλά τα πράγματα, αλλά πρέπει να τα λέμε το όνομά του. Σε ποιο κράτος ε, πάνε οι Κορεάτες και ποιε είναι οι εταιρείε που του προσλαμβάνουν. Et via quelle agence intérimaire και αυτά τα γραφεία βρέσος ε, εργασίας. Πού είναι? It, πλοκο um, uh, Πολύπλοκο είναι το σχήμα. Έχουμε ένα βορειοκορεατι έχουμε μάλλον μια κοινοπραξία που προσλαμβάνει τους ανθρώπους έπειτα κατά κάποιο τρόπο δανείζει σε αυτά τα γραφεία ευρέσου προσωρινής εργασίας πολύ μικρές εταιρείες. Και μετά πηγαίνουν σε κάποια άλλη εταιρεία και εργάζονται. Ας πούμε το ναυπηγείο στο χαρτί δεν του πληρώνει του εργαζόμενου. αλλά την εταιρεία, το γραφείο βρέσεω εργασία που τους προσέλαβε και τους έστειλε στο ναυπηγείο. Δεν είναι δηλαδή αυτή του ναυπηγείου η υπεύθυνη. Και μετά, άμα πάτε σε αυτό το γραφείο ευρέσεως εργασία θα σα πούν ότι η αρχική κοινοπραξία έφερε αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα. Πρέπει να γνωρίσετε ένα νομικό να σας απαντήσει. Είναι η απασχόληση αυτή. Ε, η το όλο σχήμα αυτό είναι εικονικό. Νομίζω είναι μια ερώτηση που μόνο ένας ε, νομομαθής μπορεί να την απαντήσει. Tout à fait, tout le débat de comment Μα ε, αυτό είναι όλο το θέμα. Πώς ο διατάκτης και όχι υπεργολάβος, ε, πρώτος, δεύτερος, τρίτος ε, είναι αυτός που έχει την ευθύνη. Λοιπόν, τώρα για 10 λεπτά η κυρία Ουταέγγι, κάπως έτσι λέγεται, υπεύθυνη εκπαίδευση από τις Κομισιόνες Ομπρέρας της Ισπανίας, του Ισπανικού Συνδικάτου. Buenas tardes a todos. Καλησπέρα σας. Ε, καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε να συμμετέχω σε αυτή την συνεδρίαση. Να πω καταρχάς, και πριν περάσω στις συνθήκες εργασίας για τους τομείς που αριστερώνουν υψηλό κίνδυνο εκμετάλλευσης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ένα πλαίσιο ε, αρχικά για να καταλάβετε με μεγαλύτερη σαφήνεια ε, τι ε, λέμε όταν μιλάμε για κάποιους ε, τομείς συγκεκριμένου δεδομένων των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και των αυστηρών πολιτικών λιτότητας που άσκησαν μεγάλες πιέσεις στους εργαζομένους λόγω του υψηλού ποσοστού Ανέργεια και της δυσκολίας αναζήτησης ε, εργασίας ή του φόβου να τη χάσουν. Δυστυχώς όλα αυτά οδήγησαν σε μια γενική επιδείνωση συνθήκες εργασίας για πολλούς εργαζόμενους που, ιδίως αυτούς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι ε, σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, κυρίως με τις την υποτίμηση που είδαμε τα δέκα τελευταία χρόνια και την προοδευτική αύξηση ανεργία. Ε, σίγουρα δεν υπάρχουν ομοιόμορφε επιπτώσει από την κρίση παντού. Υπάρχουν όμω κάποια χαρακτηριστικά, κάποια προφίλ τα οποία είναι λίγο πολύ ε, γενικά. Έχουμε του μετανάστες, τους ανέργους, μεγάλης διάρκειας, ε, γυναίκες, νέου και Μισθωτή με χαμηλή εξειδίκευση. Πρέπει να πω επίσης ότι το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών με βάση όλου τους δείκτες για το φίλο τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση αυτού του χάσματος. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει γυναικείο πρόσωπο στις περισσότερους, περισσότερες ομάδες που, είναι, ε, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκμετάλλευσης. Επίση έχουμε τους φροντιστές, ε, έχουμε τους ε, τηλεφωνητές, εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές και υπηρεσίες εστίασης, καθαριστήριες, κατοίκων φροντίδα, οικιακή βοηθή κτλ. Αυτά είναι κυρίως τα επαγγέλματα. Ε, και βλέπουμε επίσης ότι η αγοραστική δύναμη, η μισθή των ανθρώπων που είναι στη, γάτο στη βάση της πυραμίδας ό,τι αφορά τους μισθούς, ε, μέσα σε 10 χρόνια έχει χαθεί ε, το 25% της αγοραστικής δύναμης. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτά είναι πραγματικά κοφαντικά στοιχεία. Και μιλάμε και για 27% των μισθωτών για την Ισπανία που είναι στο υψηλότερο ε, βάθρο σε ό,τι αφορά την εποχικότητα των εργαζομένων. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια εποχικότητα αντίστοιχη με το 14% διπλή εμείς στην Ισπανία. Σίγουρα υπάρχει διαφορετική παραγωγική δομή και αυτό μπορεί να επηρεάσει, αλλά όχι πια και τόσο πολύ. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για τη σύντομη διάρκεια των συμβάσεων. 12 ημέρες έχει μειωθεί από το 11 έως το 16 η μέση διάρκεια. Μέση διάρκεια των συμβάσεων, εποχικών συμβάσεων, είναι 50 ημέρες τώρα. Επομένως, η επισφάλεια ουσιαστικά επηρεάζει όλους, ε, του, όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής δομής της κοινωνίας μας ε, που επιδεινώνεται λόγω των ε, ρηγμάτων και στο κράτος πρόνοιας η ευαλωτότητα αυτή, η κοινωνική, βλέπουμε να επεκτείνεται πολύ γρήγορα και να καταλαμβάνει νέους κοινωνικο-οικονομικούς χώρους, στην πρώην μεσαία τάξη όπως τη λέγαμε, όπου πλέον βλέπουμε να ε, εμφανίζονται νέα προφίλ, ε, όπως και σε πιο εξειδικευμένε θέσει εργασία, όπως είναι πληροφορική και πολιτική, μηχανική και άλλη ε, μηχανική, μηχανολόγη. Επίσης θέλω να τονίσω ότι ένα από ε, τα αίτια της ε, ε, κατάστασης είναι ότι άλλαξε η θεσμική αρχιτεκτονική στο δικό μας πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων με συνεχείς μεταρρυθμίσεις εργασιακές είδαμε να υπάρχει σημαντική επιδείνωση και ιδίως στο μοντέλο συλλογικής διαπραγμάτευσης που υποτίθεται θα έπρεπε να ρυθμίζει τις παραγωγικές σχέσεις. Με τρεις τρόπους έγινε αυτό. Απλούστε στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση και πολλαπλησιασμό στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να μην εφαρμόσει ε, τα όσα προβλέπει η συλλογική σύμβαση. Δεύτερο τρόπο είναι ε, κάποιε συλλογικέ συμβάσει εργασία που έπαψαν να ισχύουν. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα ε, στην εφαρμογή των ε, ρυθμίσεων από την εταιρεία συγκεκριμένα. Δηλαδή γίνεται μία κατά περίπτωση συνεννόηση και διαπραγμάτευση. Ε, Επομένω, έχουμε πολλές υπηρεσίες, πολλαπλών υπηρεσιών με κοινό παρονομαστή ε, την ε, μείωση, την υποβάθμιση των εργασιακών συνθήκων, ε, των μισθολογικών όρων σε σχέση με αυτά τα οποία θα είχαν συμφωνηθεί σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων με μια συλλογική σύμβαση. Κυρίως ξενοδοχικές επιχειρήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. γιατί στην Ισπανία εκεί εργάζονται πάρα πολλοί τέτοιοι εποχιακοί εργαζόμενοι. Έχουν υποδεινωθεί οι συνθήκες εργασίας τους πλέον και ουσιαστικά η κατάστασή τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ε, εκμετάλλευση. Και υπάρχει και το outsourcing, η εξωτερική ανάθεση, μια τεχνική οργάνωση και διαχείριση ε, της επιχείρησης. Στα προηγούμενα μοντέλα επιχειρήσεων υπήρχε εξωτερική ανάθεση κάποιων υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες. Καθαριότητα ή υπηρεσίες. Τώρα όμως βλέπουμε ε, να έχουμε εξωτερική ανάθεση κεντρικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης που είναι στο ίδιο το πυρήνα της εργασία μια επιχείρησης, όπως είναι το μάρκετινγκ, τα οικονομικά κτλ. Αυτές οι σχέσεις εξωτερική ανάθεσης διατηρούσαν βέβαια και κάποιο πλαίσιο πίστηση ή τέλος πάντων πλαισίωσης, γιατί υπήρχε Ήξερε και αλλά υπήρχε και μια σύμβαση που προέβλεπε ότι έπρεπε να πληρούνται κάποιοι όροι για κάποιε προποθέσει για αυτού του εργαζομένου του οποίους παλιότερα απασχολούσε η βασική επιχείρηση. Όταν φτάσαν αυτές οι, πυρε... οι εταιρείε πολλαπλών υπηρεσιών που ε, συνδέονται άμεσα με την εποχική εργασία, παρέχουν πλέον πολλές υπηρεσίες διαφορετικές και σε ένα συγκεκριμένο κλάδο αλλά γενικώ στην αγορά. Πολλαπλασιάζονται αυτές οι εταιρείες πολλαπλών υπηρεσιών. Αυτό οδηγεί σε μια διπλή πρακτική. Δεν εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις πλέον οι εταιρείε και εφαρμόζουν ε, κατά περίπτωση, ε, συνάπτουν κατά περίπτωση συμβάσει με τον εργαζόμενο σε επίπεδο επιχείρηση. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζομένων στην Ισπανία υπολογίζεται ότι δεν προ, ε, καλύπτονται πλέον από συλλογική σύμβαση εργασία και αυτό έγινε μέσα σε 6 χρόνια. Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτών των επιχειρήσεων πολλαπλών υπηρεσιών μέχρι στιγμή είναι ακριβώ ότι δεν μπαίνουν, δεν ταιριάζουν στο μοντέλο συλλογική διαπραγματεύση που, έχει σχεδιάσει, που έχουν σχεδιαστεί με βάση του κανόνε που ίσχυαν. Και οι περισσότερε από αυτέ τι επιχειρήσει δεν εφαρμόζουν καμία σύμβαση. Το επόμενο ε, βήμα είναι η διαπραγμάτευση της σύμβασης από την ίδια την επιχείρηση με προτεραιότητα. Έτσι μπορούν να διαπραγματευτούν τις δικές τους συμβάσεις με το προσωπικό. Και έτσι μειώνεται και ε, υποβαθμίζονται οι συνθήκες εργασίας και ιδίω οι μισθολογικοί όροι. Είχαν αυτές οι, τα γραφεία βρέσου εργασίας επίσης. Μέχρι 8 χρόνια πριν αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να εφαρμόζουν τους ίδιους όρους με τη βασική επιχείρηση. Υπάρχει ένα κενό με αυτές τις νέες εταιρείε ε, πολλαπλών υπηρεσιών που ακριβώς βοηθά στο να μην τηρούν ούτε καν αυτούς τους όρους και αυτές τις προϋποθέσεις που ίσχυαν για τα γραφεία βρέσεως εργασίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να να ανατραπεί αυτό το μοντέλο με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ε, προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να βλέπουμε αύξηση των κερδών της επιχείρησης και τελμάτωση των μισθών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μην ανησυχείτε. Αριστερά σας είναι η βοηθή των πολιτικών ομάδων που καταγράφουν προσεκτικά αυτά που είπατε και τα οποία θα τα μεταφέρουν έστω και δεν υπάρχουν εδώ βουλευτέ. Και δεξιά έχετε του εκπροσώπου τη Κομισιόν, που και αυτοί ακούν προσεκτικά αυτά που λέτε και πώς σας λένε σας είπαμε ε, κάποιος από εσά έγραψε τέλο πάντων την οδηγία, ήταν του συντάκτη τη οδηγία για του αποσπασμένου. Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή η εκμετάλλευση δεν σταματά στην ε, απόσπαση των εργαζομένων. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει. Εγώ πάντω θα κάνω μια παρατήρηση. Αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτά που είπατε ήταν η εκμετάλλευση των γυναικών σε όλου του τομεί. Αυτό που δείχνει βέβαια το ότι οι γυναίκε όταν δουλεύουν. Α, καλωσόμουν κυρία Κωνσταντιέ, η οποία ήταν συνσυντάκτη στην οδηγία για του αποσπασμένου. Έχουμε λοιπόν μια οργανωμένη ανασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν της νομοθεσίας που διέπει την ε, μετακίνηση των εργαζομένων. Αυτούς παρατήρηση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ε, συγκεκριμένες θέσεις. Η εκμετάλλευση των γυναικών είναι κάτι το οποίο με τρομοκρατεί πραγματικά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Χαίρομαι γιατί η εξειδίκευσή μου η επαγγελματική μία από αυτές αφορά την ανάλυση των συνδικών ισότητας που αφορά τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη όλων αυτών των πτυχών που στο εσωτερικό των επιχειρήσεων επιτρέπει την ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ όλων ώστε να εφαρμόζεται αρχή της ισότητας τη επιχειρήση. Αυτό ανάγεται στο 2007 στην Ομοθεσία για την ισότητα που έχουμε εμείς. Όπως έλεγα στην αρχή, είχαμε και την οικονομική κρίση και έχουμε τις ιδεολογικές αρχές που διέπουν την κοινωνία στην οποία ζούμε. Και γι' αυτούς τους λόγους το θέμα αυτό έμεινε σε δεύτερο πλάνο σε σχέση με άλλα θέματα προτεραιότητας. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια πάντως ότι όλοι οι δείκτες της αγοράς εργασίας, όλοι οι δείκτες της αγοράς εργασίας ε, περιλαμβάνουν μια συνιστόσα φύλου και εξηγούν ακριβώς την θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας. Οπότε, αν θέλετε, μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να μιλήσουμε για περιπτώσεις που εκεί όπου υπάρχει πραγματική εκμετάλλευση είναι κάτι που αφορά τις γυναίκες. Αν δεν ήταν γυναίκες, αυτοί οι εκμεταλλευόμενοι, η νομοθεσία θα είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά παραδοσιακά αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες γινόταν ας πούμε στο σπίτι με τη θέση της γυναίκας στο σπίτι αφορά αυτό που ονομάζουμε σήμερα το χάσμα, το φιλετικό. Τη διαφορά δηλαδή στις συνθήκες ισότητας μεταξύ άντρων και γυναικών. Αυτά προς το παρόν. Αν θέλετε κάτι άλλο μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Τώρα για 10 λεπτά. Ο λόγος του κύριου Ντέρινγκ υπεύθυνο ποινικού δικαίου από την Υπηρεσία Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Βιέννης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Sorry. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη δουλειά μας. Είναι ένα θέμα που αφορά τους πάντες παρά τις απουσίες που έχουμε σήμερα. Εμείς κάναμε έρευνα σε σχέση με τις ε, ακραίες περιπτώσεις εκμετάλλευσης εδώ και πέντε χρόνια. Θα το συνδυάσω αυτό με αυτό που ονομάζουμε Selex, δηλαδή σοβαρές μορφές, ακραίες μορφές, εγκληματικές μορφές εκμετάλλευσης. Δηλαδή μορφές οι οποίες είναι στην ουσία επαρκείς για να θεωρηθούν ποινικέ στις χώρες μέλη. Αυτό εξετάζαμε λοιπόν εδώ και κάποια χρόνια. Υπάρχει βέβαια μια νοτική νομική συγγνώμη, βάση, χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπου έχουμε την απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας και η επιβολή αποδεκτών συνθηκών εργασίας. Παράγω δίκαιο. Υπάρχει μεγάλο παράγωγο δίκαιο σχέση με αυτό το θέμα. Δικαιώματα των θυμάτων και αυτό αφορά διάφορους τομείς. Δηλαδή η νομοθεσία για το και εργασία κτλ. Για μας αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό είναι η οδηγία που αφορά τους εργοδότες, την εργοδοσία, γιατί αυτό επιβάλλει στις χώρες μέλη να δράσουν κατά κάποιων μορφών εκμετάλλευσης. Και υπάρχει ένας ορισμός εδώ. Οι ακραίες μορφές εκμετάλλευσης. Και αυτό σχετίζεται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλαδή, μορφές εκμετάλλευσης που σχετίζονται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έχουμε και αυτή την έκθεση, που ήταν η πρώτη έκθεση που αφορούσε την εκμετάλλευση, και που βασίζεται σε 660 συνεντεύξεις επαγγελματιών και συζητήσεων και με κάποιες ε, περιπτώσεις που αφορούν διάφορους τομείς της, οικονομίας. 27. Με μια ποικιλομορφία καταστάσεων που εξετάσαμε. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω από την αρχή είναι το εξή. Ίσως το κύριο πρόβλημα που ισχύει εδώ είναι η ατιμορρησία. Δηλαδή, οι ακραίες μορφές εκμετάλλευσης, ποινικής μορφής, λαμβάνουν χώρα χωρίς να γίνεται τίποτα. Και ο λόγος αυτής της ατιμορρησίας είναι κυρίως τρεις που αναφέρουμε εδώ στην διαφάνεια έλλειψη εποπτείας, έλλειψη ενεργού διερεύνηση εκ μέρους αστυνομίας και έλλειψη υποστήριξης των θυμάτων. Δηλαδή τα θύματα δεν ενθαρρύνονται να απευθυνθούν στην αστυνομία. Στην πρώτη έκθεσή μας τονίσαμε και υπογραμμίσαμε τομείς που είναι επιρρεπείς στην εκμετάλλευση, γεωργία καταρχάς, δασοκομεία, αλληλεία, κατασκευές, βιομηχανία, ξενοδοχεία, διατροφή, τρόφιμα δηλαδή, οικιακές βοηθή, μεταποίηση τροφίμων, που είχαν εξέχουσα θέση στις μελέτες μας. Εδώ λοιπόν καταγράφουμε κάποιες από τις περιπτώσεις όπου βρήκαμε περιπτώσεις εντό εκμετάλλευση. Ολοκληρώνουμε τώρα το δεύτερο γύρο έρευνών μας που θα οδηγήσει σε τρεις δημοσιεύσεις. Η πρώτη για τις οικιακές βοηθούς, τους οικιακούς βοηθούς, έχει ήδη διανεμηθεί ηλεκτρονικά. Στη δεύτερη έκθεση μιλάμε για το πώς γίνονται πώς γίνεται η εποπτεία στο χώρο της εργασίας. Αυτό θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβρη και μετά έχουμε μια μεγάλη συγκριτική έκθεση που θα δημοσιευθεί στο πρώτο μισή του χρόνου. Στην έρευνά μας είχαμε συνεντεύξεις με εργαζόμενους αποκλειστικά. Αυτή, σε αυτή τη φάση είχαμε λοιπόν μόνο εργαζόμενους και οι πρώτες έρευνες μας αφορούσαν τους γειακούς βοηθούς. Είχαμε 51 συνεντεύξεις με περιπτώσεις εκμετάλλευσης ατόμων που δουλεύαν ως οικιακή βοηθή. Οι χώρες που καλύπτονται στο δεύτερο γύρο της έρευνάς μας στον πρώτο γύρο είχαμε 21 χώρε, στο δεύτερο γύρο είχαμε 8. Όπως λέγαμε, ο δεύτερο γύρο ερευνών αφορά συνεντεύξεις εκμεταλλευόμενων εργαζομένων εποχιακούς, γεωργικούς βοηθούς, διανομής, Στην Ένωση έχουμε και περιπτώσει εργασιακή μετανάστευση, α πούμε, από τη Βουλγαρία στη Γαλλία ή από την Πολωνία στην Ιρλανδία. Εντό Ένωση δηλαδή, που λάβαμε υπόψη μα. Και οι συνεντεύξει μα ε, αυτέ αφορούσαν σε περιπτώσει εκμετάλλευση από το 2013 μέχρι το 2018. Βλέπετε και ένα χάρτη που αφορά την καταγωγή των εργαζομένων και τονίζει ακριβώ τι ε, περιπτώσει εκμετάλλευση από νέε χώρε μέλη, εργαζομένων από νέε χώρε μέλη. Στόχευσή μα είναι να εντοπίσουμε παράγοντες κινδύνου ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που οδηγούν στην εκμετάλλευση. Αυτό σχετίζεται με το πώς ακριβώς γίνονται οι επιθεωρήσεις εργασίας ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Είχαμε συνεντεύξεις επίσης εργαζομένων όπου του ζητήσαμε να μας πούν τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά κατά την άποψή τους σε σχέση δηλαδή με την προσφυγή στην αστυνομία ή γενικά με την δημοσίευση των σπάδων των περιπεντιών τους. Είχαμε μια πρώτη δημοσίευση μόλις τώρα την Παρασκευή σε σχέση με τους οικιακούς βοηθούς. Εκεί είδαμε ότι για αυτές τις περιπτώσεις είχαμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις εκμετάλλευσης, το οποίο σημαίνει ότι από τους 51 εργαζόμενου που είχαμε συνέντευξη για αυτό το τομέα, πάρα πολλοί είχαν δεχτεί συμπεριφορά η οποία παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πολύ συγκεκριμένε μορφές ε, όπως ε, σεξουαλική παρενόχληση, φυσική βία, η εργασιακή εκμετάλλευση δεν αφορά μόνο την καταγκαστική εργασία. Έχουμε περιπτώσεις βίας και στις περιπτώσεις των γιακών βοηθών έχουμε αυτές τις ε, μορφές εκμετάλλευσης. Έχουμε επίσης και περίοδους για τις οποίες είναι απλήρωτοι, πολύ χαμηλή αμοιβή. Αυτό το βρήκαμε βέβαια να ισχύει σε όλους τους τομείς της εκμετάλλευση, ιδιαίτερα για τις υπερορίες και την ε, αμοιβή η οποία δεν ήταν κατάλληλη. Αλλά είναι πιο έντονο αυτό το θέμα με τους οικιακούς βοηθούς, όπου έχουμε πλήρη έλεγχο ή εξάρτηση των εργαζομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνια. Δεν κάνουμε μόνο έρευνα λοιπόν, αλλά και παρέχουμε συμβουλές και αναζητούμε λύσεις. Να παρθυμίσω κάποια απλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ας πούμε, είδαμε ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας ήταν επαρχής. Το είπαμε ήδη δύο φορές βέβαια. Ένα βήμα πρόοδου θα ήταν να επικυρώσουν όλες οι χώρες μέλη τη σύμβαση για τους σχιακούς βοηθούς. ώστε να δοθεί άδεια για επιθεωρήσεις εργασίας. Δεν ξέρω στις χώρες μέλη ποιος κάνει αυτό το είδο επιθεώρησης εργασίας ή δεν ξέρω κατά πόσο έχουν την δικαιοδοσία να μπουν σε αυτά τα σπίτια και να επιθεωρήσουν αυτές τις μορφές εργασία αν έχουν βέβαια την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του σπιτιού ή του διαμερίσματος. Ως παράγοντας κινδύνου, επίσης είναι η του διαμερισματο ως παραγοντα κινδυνου επισης ειναι η προσβαση στην στήριξη. Θα πρέπει να στοχεύσουμε εδώ στις υπηρεσίε στήριξη, και αυτό ισχύει και για άλλε μορφέ ε, μορφές ε, εγκλημάτων, σεξουαλική παρενόχληση παιδιών, η εκμετάλλευση. Παρ' όλα αυτά είναι περίπλοκο εδώ το ζήτημα και νομικά αλλά και πρακτικά γιατί σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλά καταρτισμένους και καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους για την παροχή στήριξης σε αυτόν τον τομέα. Ένας παράγοντας κινδύνου είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, δεν γνωρίζουν ποιον να απευθυνθούν και πώς να πληροφορηθούν. Οπότε το να αυξήσουμε την επίγνωση, τη συνειδητοποίηση αυτών των εργαζομένων για τα δικαιώματά του. θα ήταν σημαντικό βήμα μπροστά. Θα καταλήξω, γιατί ήδη έχω περάσει το χρόνο μου. Ναι, βεβαίω οι εργαζόμενοι σε κάποιες σε κάποιους οικονομικούς τομείς έχουν ψηλότερο κίνδυνο εκμετάλλευση. Ανέφερα του οικιακού ε, βοηθού ένα από του κυριότερου κινδύνου. Αλλά νομίζω ότι οι απαντήσει μα θα πρέπει να εγγράφονται στο δίκαιο, λαμβάνοντα υπόψη μια περίπλοκη νομοθετική κατάσταση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αυτά που ξέρουμε πρακτικά και εμπειρικά. Να λάβουμε υπόψη μα και τι συμβουλέ ε, εμπειρογνωμόνων και των ίδιων των θυμάτων. Στόχος μας είναι εδώ να επιτρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς να μιλήσουν, να πάνε στην αστυνομία και να δικαιωθούν μέσω προσφυγής δικαιοσύνη, αποσημείωση κτλ. Πρέπει λοιπόν καταρχάς να πετύχουμε την πρόσβαση αυτών των ατόμων στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε κυρία Ντέρινγκ. Θα Πρέπει να δώσω τη θέση μου στην κυρία Τζέα να αναλάβει την Προεδρία. Αν υπάρχουν βουλευτέ που έχουν ερωτήσεις, παρακαλώ, καλούνται να πάρουν το λόγο. Όσο μας είπατε, είναι πολύ ανησυχητικά. με ανησύχησε πάρα πολύ αυτές οι σοβαρές παραβιάσεις και η ατιμορρησία και μας ε, δώσετε και ένα ορισμό των πληγέντων τομέων. Μιλήσατε και για τα κράτη-μέλη. Όμως ε, αυτό αφορά περισσότερο τα κράτη στη Δύση προς την Ανατολή και αναφερθήκατε ε, στο πάνελ. Έχω μια αμφιβολία σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων ε, που ρωτήθηκαν και πώς μπορείτε να μας αναφέρετε και κάποια πληροφορίες για τα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, ε, αναφέρομαι όσα είπε ο κύριος Μπρούκερ, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας να μπορεί αποτελεσματικά να παρέμβει. Η Κομισιόν θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Η επιθεώρηση εργασίας έχει λίγα μέσα, αλλά πώς μπορούμε να τους εξοπλίσουμε με περισσότερα μέσα. Θα σας ακούσω και μετά θα φύγω. Να απαντήσω ναι, φυσικά η επιθεώρηση στον τόπο εργασία ε, είναι το κυριότερο. Πρέπει οι επιθεωρήσει αυτέ να λειτουργήσουν. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πρώτο βήμα, δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Το Σεπτέμβριο θα δημοσιεύσουμε μία μικρή έκθεση που θα αφορά μόνο πώς να οργανώσουμε τις επιθεωρήσεις επιτόπου στο χώρο εργασίας έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και εγκληματικές ε, καταστάσεις, εγκληματικές μορφές ε, εκμετάλλευσης ε, όπου θα πρέπει να δοθεί κάποια συνέχεια. Φυσικά πρέπει να υπάρχει συνεργασία και μεταξύ αστυνομία, εισαγγελέων και επιθεώρησης εργασίας. Αυτό έχει να κάνει με το πώς οργανώνονται αυτοί οι συσχέτιση, αυτός ο συσχετισμός μεταξύ των δημοσίων αρχών. Λάουρα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τζουζέπε Ιουλιάνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω την μητρική μας γλώσσα τα Ιταλικά. Καθώς δίνεται η δυνατότητα. Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία γιατί φυσικά η δική σας παρέμβαση ουσιαστικά επισέρχεται σε όλο αυτό τον προβληματισμό που κάνουμε για το θέμα της ε, εκμετάλλευσης. Εμείς ε, έχουμε υλοποιήσει πολύ συγκεκριμένες ε, γνωμοδοτήσεις για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως θέλω να προσπαθήσω να κάνω μια παρέμβαση που να αρμόζει στο πλαίσιο. Όπως είπαν οι προλαλήσατες, αναφέρουμε και στη συνάδελφο Μαγιατόγουαϊ από τις Κομισιόνες Ομπρέρας και εγώ προέρχομαι από τα συνδικάτα. Ξέρετε ότι η κοινωνική, στην Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή συμμετέχουν ε, και οι επιχειρηματίες ε, αλλά ε, και τα συνδικάτα και άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για ανθρώπους που ούτως ή άλλως έρχονται σε επαφή με αυτό το φαινόμενο της καταναγκαστικής εργασίας. Και πράγματι, ίσως να μην έχουμε μεγάλη παρουσία βολευτών αυτή τη στιγμή, όμως ε, σίγουρα θα δοθεί συνέχεια από όσους συμμετέχουμε στη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω να υπάρχει ισχυρή συμμαχία, κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να δοθεί όθηση σε αυτά τα θέματα που συζητούμε και για να υποστηριχτεί διαλεκτική το διαλεκτικό αλλά και το συμβουλευτικό έργο που κάνουμε εμείς ως ΕΟΚΕ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς αναγνωρίζεται ο ισχυρός ρόλος των κινητήριων δυνάμεων της οικονομίας, γιατί και εμείς θυγόμαστε. Το να μιλάμε σήμερα για καταναγκαστική εργασία είναι κάτι παράλογο. Αλλά γιατί μιλάμε, γιατί εμείς θέτουμε στο επίκεντρο ε, πάντοτε την ε, παραπομπή στις διεθνείς συμβάσεις της ΔΟΕ. Αλλά όπως ε, ξέρετε, υπαριθμόν 29 και 105 συμβάσεις ακριβώς αναφέρονται στην καταναγκαστική εργασία. Μία είναι του 1995 και η άλλη του 1957. Όταν γινόταν αναφορά στην καταναγκαστική εργασία, ως αντικείμενο των κρατών. Δηλαδή, όταν τα κράτη ασκούσαν καταναγκαστική εργασία. Τώρα, τι συνέβη μετά. Επικεντρωνόμαστε στην ιδιωτική οικονομία και η καταναγκαστική εργασία λόγω της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης, της ε, παραοικονομίας ε, διαδίδεται και τα εγκληματικά δίκτυα παίρνουν ε, τεράστιες διαστάσεις και αυτό αφορά και την ε, δική μας, την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Εμείς ε, υλοποίησαμε μια γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν, το τμήμα ΡΕΚ, εξωτερικής πολιτικής, την 395 γνωμοδότηση. Και αρκεί να αναφέρετε αυτά τα στοιχεία και φυσικά θα έχετε πλήρη τεκμηρίωση. Όμως ήθελα να κάνω κάποια σχόλια εμείς. Αυτό το πρόβλημα των συνθήκων που είναι θεμελιώδης το έχουμε θίξει και μέσω της γνωμοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2011 να μπορεί να γίνει ένα είδος πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ε, σύμβαση του 99 για να αντιμετωπίσουν παραδείγματος χάρη την εμπορία ανθρώπων καθώς ε, υπάρχουν πολλά κενά ως προς την προστασία των θυμάτων, την ε, πρόληψη, την ε, τιμωρία των διακινητών. Πρέπει να πάρουμε κάποιες διατάξεις που υπάρχουν σήμερα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι ζωτικές δυνάμεις της οικονομίας έχουν κάνει αυτήν την έκκληση και ουσιαστικά αν την υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει πολύ μεγάλη δυναμική. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος στόχος της συζήτηση σήμερα, γιατί αν ε, οι θέσεις αυτές υιοθετηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την ε, Κομισιόν, τότε θα πάμε εμείς ε, πέρα από το συμβουλευτικό μας ρόλο σε ΟΚΕ. Εμείς αυτές τις μέρες συζητάμε για τη βιομηχανία 4.0. Ο υπουργό Σόιμπλε τρομοκρατεί του συμμετέχοντες στον Ταβός όταν μιλά για 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάρη στη βιομηχανία 4 αλλά και την ε, απώλεια 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Αν προσθέσουμε τα δύο και αφαιρέσουμε τα, τα μιλάμε για 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, που χάνονται και αυτό έχει τρομοκρατήσει τώρα επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτά είναι τα νούμερα, εγώ συνδικαλιστής ε, σας λέω ότι Λυπάμαι όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε 185 εκατομμύρια παιδιά που σήμερα δουλεύουν. 80 εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες ε, και εμείς ε, ουσιαστικά μιλάμε για σκλαβιά εδώ και δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχουν. Μιλάμε για δήλωτη εργασία, αλλά μιλάμε για σκλαβιά. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι πολύ ζωτικό γιατί αφορά τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς ή να κάνουμε απλώς ε, μια ακαδημαϊκή συζήτηση εδώ. Εμείς έχουμε κάνει αυτές τις προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις φτάνουν στην ε, Κομισιόν. Κάθε έξι μήνες έρχεται μια μελέτη στην ΕΟΚΙ και αναφέρονται διάφορα στοιχεία που έχουν υιοθετηθεί, όμως δεν αρκεί να λέμε ότι το 80% των γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ στη συνέχεια θετούνται έχουμε και το θέμα της εφαρμογής που ουσιαστικά εξαρτάται αν υπάρχει πολιτική πρωτοβουλία. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε διάφορες γνωμοδοτήσεις για την κατεστική εργασία, για την παραοικονομία, για την αδήλωτη εργασία, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών, για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, για την ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την κοινωνική συμμετοχή, στην συνεργασία και στην ανάπτυξη. Όμως λείπει μια συνοχή μεταξύ όλων αυτών των πολιτικών. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν υπάρχει ισχυρή πολιτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να μιλάμε για την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη, για τη δέωση επιμέλεια, πολύ ωραία. Αλλά όταν ε, οι μεταναστευτικές πολιτικές ε, ε, δεν προκρίνουν αλλαγέ. Όταν ε, τα αιτήματα που κάνουμε εμείς στα κράτη δεν ε, εισακούονται, βρισκόμαστε μπροστά σε έκρηξη πολύ ενισχυτικών φαινομένων. Έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, με την ίδια την επιβίωσή του. Ζητώ συγγνώμη αν μίλησα κάπως πιο συναισθηματικά, όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό Ε, η πρόεδρος είπε ότι ζητά συγγνώμη για κάποιες απουσίες. Ε, πραγματικά ε, με συγκίνησε. Όμως όλα τα δεδομένα που αναφέρονται εδώ θα διαβαστούν γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή δράση πολιτική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Ιουλιάνο. Τώρα. Αν ε, θέλουν κάποιοι συνάδελφοι το λόγο, μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Βάσει και των ε, όσων μας είπατε και των δεδομένων που μας δώσατε. Και ακούσαμε και κάποιες προτάσεις που ίσως θα πρέπει να υιοθετήσουμε όταν ε, θα λειτουργούμε ως συνομοθέτες. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη φιλοδοξία, ίσως κάνουμε, γιατί πολύ συχνά έχουμε δει τι συμβαίνει στους τριμερείς διαλόγους. Πολύ συχνά μπορεί να δοθεί μια ενίσχυση ακόμη και μέσα της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μωρέν Σαρτιά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για την ακρόαση. Και θέλω να πω πως με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχω ασχοληθεί με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ανησυχώ γιατί πραγματικά δεν έχουμε στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε μερικά στοιχεία, ελλειπή. Δεν ξέρουμε όμως ε, ε, πώς η εργασία κρυφή, αν θέλετε, υπάρχει. Δηλαδή μόνο ένα κομμάτι του παγόβων βλέπουμε. Αν θέλουμε να αντιδράσουμε ε, πολιτικής πλευράς θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ πιο βαθιά και να αναλύσουμε την πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ή γενικά χαρακτηριστικά είχαμε, αλλά δεν βλέπαμε τι γίνεται στην πραγματικότητα και ποιο είναι το εύρος της κατάστασης. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκής ε, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να δούμε πώς έχει πραγματικότητα. Και η κατοίκον εργασία δεν επιτρέπει να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα ήταν πάρα πολύ σημαντικά για να προχωρήσουμε σε μια πολιτική αντίδραση. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όλοι μαζί για αυτά τα δεδομένα, τα κρυφά, για να βγουν στο φως και να προκαλέσουν την πολιτική αντίδραση που εσείς περιμένετε, κύριε Τζουλιάν. Δεύτερο, με πολύ μεγάλη προσοχή άκουσα τα περιφύλου. Να σας πω πώς το βλέπουμε εμείς, το θέμα του φίλου σε επίπεδο κρατών, μελών, σε επίπεδο οικογενειών και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κάνουμε πολλά για να έχουμε την ε, ίση, ίσες ευκαιρίες και ισότιμη εκπαίδευση ε, ανδρών και γυναικών. Ε, τα ποσοστά είναι 60% γυναίκες με δίπλωμα. Αν δούμε τις γυναίκες που είναι θύματα στο που αναφέρατε, εδώ έχουμε αντιστροφή και πολύ περισσότερο αυτού του λόγου άνδρες-γυναίκες. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την επιτυχία των γυναικών στην εκπαίδευση και δεν αντικατοπτρίζεται αυτό ε, στην επιτυχία αντίστοιχη των γυναικών στον ε, ε, χώρο εργασίας. Είναι αντίστροφα τα ποσοστά, αντιστρόφως ανάλογα. Και δεν πρέπει να μην είναι έτσι τα πράγματα. Για να μιλήσω για την κατοίκον εργασία, οι γυναίκες είναι αυτές που είναι και τα μεγαλύτερα θύματα. Θέλω να μιλήσω και για το πρόβλημα των παιδιών. Παιδική εργασία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Μας δώσατε κάποια στοιχεία για 80 εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται. Πράγματι. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ποια είναι η πραγματικότητα. Λέτε 80 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται. Εμείς μέσα μας λένε ναι, αλλού. Όχι εδώ στην Ευρώπη, αλλού. Αυτό είναι πάλι το θέμα, να έρθουμε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, να δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα. Δεν το ξέρουμε και όσο δεν το ξέρουμε δεν θα υπάρξει πολιτική αντίδραση. Αν δεν νιώσουμε ντροπή μπροστά στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να αντιδράσουμε. Το τρίτο σημείο. Επειδή είναι κρυμμένα όλα αυτά, κρυφό το σύστημα. Δεν υπάρχει προστασία. Μπορεί να προβλέπονται κάποιες δυνατότητες στο δίκαιο των κρατών μελών, αλλά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν ε, την προστασία αυτή που θα τους παρέχει δικαιοσύνη, το κράτος κτλ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κανείς που να μένει στο απειρόβλητο από το κοινωνικό ιστό. Alors, oui, du Θεώρηση εργασίας, μάλιστα, ναι. Όμως, ξέρετε, η θεώρηση εργασίας, ε, συμφωνώ, συμφωνώ, είναι αυτό που είναι. Αλλά όταν έχουμε μετακίνηση διεθνούς εργατικού δυναμικού δεν έχει δυνατότητες επιθεώρησης εργασίας να κάνει σωστά τη δουλειά της. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και δεδομένα τα οποία να διαβιβάζει τον κράτος μελωστά. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν εγώ είναι να έχουμε ε, μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, ε, να γίνει αυτή η πρόταση από την Κομισιόν. σε αυτό το τομέα βλέπουμε αμέσως ότι υπάρχει ένα σημαντικό πεδίο εργασίας που θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, δεν αρκούν οι προθέσεις για να υπάρξει πολιτική αντίδραση. Πρέπει να αντιπαραβάλλουμε την πολιτική με την πραγματικότητα. Είπατε και για τις επιχειρήσεις, ότι ισχύει το ίδιο στις επιχειρήσεις. Ναι. Υπάρχουν ρεύματα εκμετάλλευση εντός Ευρώπης. Υπερβαίνουν όμως ε, τις ε, επιχειρήσεις. Εκμεταλλεύονται κάποια κυκλώματα ε, την κατάσταση και έχουμε εκμετάλλευση Ανατολής από τη Δύση. Το βλέπουμε τους αποσπασμένους εργαζόμενους και με την κρυφή αυτή εργασία, την παραοικονομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε τα μεγάλα μέσα. Αν θέλουμε να υπάρξει πολιτική αντίδραση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Γιατί το ένα από το άλλο δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Χάβι Λόπες για πέντε λεπτά. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με τα γενικά σχολεία και την ευκαιρία που έχουμε ως Ένωση και Κοινοβούλιο να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων με την οδηγία της Κομισιόν. Όπως ξέρετε, στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε πέρυσι το φθινόπωρο υπάρχει η δυνατότητα για νέα νομοθετικά μέτρα ένα από αυτά είναι μπροστά μας για να το συζητήσουμε σήμερα το πρωί το συζητήσαμε κιόλας η οδηγία για τις συνθήκες εργασίας ευκαιρία νομίζω για να ρυθμίσουμε ως αυτές τις βλαβερές πτυχές της αγοράς εργασίας. Αβεβαιότητα, ορομίστη, νέες πλατφόρμες, ανασφάλεια δηλαδή. Θέματα που σχετίζονται με πιο σημαντικά ζητήματα όπως η αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους γενικότερα. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τι θα μπορούσε να κάνει ω συγκεκριμένη ε, πρόταση το Κοινοβούλιο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στις μήνες. Αυτό θέλω να μου πείτε. Δεύτερον, ένα από τα εργαλεία του 20ου αιώνα για την εξορρόπηση των εργασιακών σχέσεων ήταν οι συλλογικέ συμβάσεις. Αναφερθεί και η μόχλευση μέσω της αύξησης των απολαβών. Αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν εξασθενήσει οι συλλογικές συμβάσεις. Οπότε αυτό το εργαλείο που είχαμε παλιά και που χρειαζόμαστε οικονομικά, την αύξηση δηλαδή των μισθών. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο εκεί όπου δεν χρησιμοποιείται και πώς το ενισχύουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα φαινόμενα στην αγορά εργασία. Γιατί και για τον 21ο αιώνα μάλλον θα συνεχίσει να αποτελεί το κυριότερο εργαλείο. Ευχαριστώ. Το συνάδελφο Λόπες. Πριν να πω και εγώ τα δικά μου, ως μέλος της Επιτροπής, ομολογώ ότι συγκινούμε γιατί δεν μου είχε ξανασυμβεί εδώ στην Επιτροπή και θα πω και τις δικές μου παρατηρήσεις. Πάντως χαίρομαι πολύ, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που καλωσορίζω τους εκπροσώπους του Συλλόγου Τυφλών της Προβυγγίας και των συνοδευτικών σκυλιών Χαιρόμαστε που σας καλωσορίζουμε. Λέμε πάντα εδώ καλωσορίσατε στο σπίτι σας γιατί η Ευρωβουλή είναι το σπίτι των πολιτών, το σπίτι του λαού. Μετά βέβαια και η Κομισιόν θα πρέπει να μας μιλήσει. Ο Δόκτωρ Περέιρα θα λάβει το λόγο στη συνέχεια. Αλλά Επιτρέψτε μου να πω και εγώ κάποια πράγματα. Μου είναι προσφυλές το θέμα γιατί πριν από τέσσερα περίπου χρόνια όταν έφτασα στην Ευρωβουλή σε μία συνάντηση των συντονιστών ζήτησα το λόγο για ένα πρόβλημα που αφορά μορφές καταναγκαστικής εργασίας στην Ιταλία μορφές κλαβιά στην ουσία. Ήταν δύσκολο να μεταφραστεί η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς στα Ιταλικά. Και έπρεπε να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν αφορά βέβαια μόνο την Ιταλία, αλλά δυστυχώς και άλλες χώρες και συνδέεται με τον τομέα της γεωργίας στον οποίο εμπλέκονται τα περισσότερα άτομα που αντιμετωπίζουν αυτές τις μορφές σκλαβιάς αλλά όχι μόνο και αλλού και στην εστίαση, στον τουρισμό, στις ε, οικοδομές τομείς που παρουσιάζουν ψηλό επίπεδο εκμετάλλευσης. Σε αυτούς λοιπόν τους τομείς βρίσκεται η μήτρα αυτού του φαινομένου. Ιδιαίτερα στο νότο και την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού με σοβαρό αντίκτυπο και ζημιές και βλάβες στο κοινωνικό ιστό, γιατί δεν αφορά μόνο το άτομο το οποίο εκμεταλλεύονται, το οποίο είναι απλήρωτο, δεν προστατεύεται και ζει σε συνθήκες που είναι δύσκολο να διαφύγει. Αλλά αφορά γενικότερα την κοινωνία. Επειδή δημιουργείται ένας μηχανισμός όπου μαζί με την ε, πρόσληψη υπάρχουν και άλλες προβληματικές. Σήμερα τα δεδομένα μας λένε ότι η εκμετάλλευση μετατοπίζεται έντονα προς τις γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες υπόκεινται περισσότερο στην εκμετάλλευση και τη δουλεία. πορνίας ας πούμε, και εκμετάλλευση εκεί. Σήμερα έχουμε εκμετάλλευση και των ανηλίκων και των παιδιών, κυρίως στα καλοκαίρια και σε συγκεκριμένους τομείς. Η βλάβη λοιπόν η ζημιά επεκτείνεται. Και αυτοί οι τομείς δεν αντιμετωπίζουν κρίση. Αυτό πρέπει να το πω. 880.000 πολίτες υπολογίζουν σήμερα στην Ευρώπη τους ε, πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός παρουσιακών μορφών πρόσληψης χωρίς καμία εγγύηση με τζίρο 25 δις 25 δις δηλαδή είναι ο τζίρος αυτής της παρανομίας ως κύκλος εργασιών και αποτελεί μια σιωπηλή καταστροφή, ένα σιωπηλό δράμα, γιατί το συζητάμε μόνο όταν πεθαίνει κάποιος. Μια γυναίκα, ας πούμε, στις καλλιέργειες ντομάτας στο νότο, πεθαίνει από την κούραση, επειδή δεν αντέχει την καταπώνηση και τη ζέστη. Τότε μόνο συζητάμε αυτά τα θέματα. Δυστυχώ σήμερα η νομοθεσία που χρησιμοποιείται σε αυτό το κλάδο δυστυχώς δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρομακτικά στοιχεία. Υπάρχει η 51 οδηγία του 2009, τις οποίες όμως οι διατάξεις εφαρμόζονται ελάχιστα και προβλέπεται η τιμωρία του τελικού χρήστη, δηλαδή του επιχειρηματία αυτής της μορφής εκμετάλλευσης. Αλλά οι τα ίδια τα θύματα αντιμετωπίζουν αντίπεινα και απελάσεις. Έβλεπα τα στοιχεία τα οποία είναι τρομακτικά αμοιβή 20 ευρώ τη μέρα για 13-14 ώρες εργασίας. Ένα σάντουιτς το οποίο πληρώνουν αυτοί 5 ευρώ, ένα μπουκαλάκι νερό 3 ευρώ και η ενδιάμεση αυτοί που προσλαμβάνουν αυτά τα θύματα πληρώνονται από τα ίδια τα θύματα και αυτοί εκπαιταλεύονται τα θύματα με τη σειρά τους. Αυτή λοιπόν η νομοθεσία δεν αρκεί. Θα πρέπει να τιμωρήσουμε αυστηρά και τους ενδιάμεσους, αυτούς που κάνουν τις προσλήψεις. Θεσπίστηκε στην Ιταλική νομοθεσία αυτό το έγκλημα με φυλάκιση 5 έως 8 χρόνια και πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργάτη που προσλαμβάνουν. Θα πρέπει λοιπόν να παρανεύουμε περισσότερο και καλύτερα με αποτελεσματικό τρόπο, ας πούμε προβλέποντας επιθεωρήσεις διαγωνισμών που περιλαμβάνουν αδήλωτη εργασία. Θα πρέπει να έχουμε ισότητα στις αγορές, έστω και αν θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα, ξέρουμε ότι για τους εργαζόμενους είναι δύσκολο να προσφύγουν κάπου Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να παρενεύουμε με επιθεωρητέ εργασίε οι οποίοι θα είναι καλά καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι για αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά θα μπορούσαμε να παρενεύουμε και για το θέμα των γυναικών. Γιατί έχουμε ένα ανατριχιαστικό στοιχείο. Στην Γεωργία έχουμε γύρω στις 15.000 γυναίκες οι οποίες προσλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο εκμετάλλευσης. Άλλες τόσες γυναίκες είναι στο νότο. Αυτά τα στοιχεία δεν επιδέχονται ερμηνεία. Απαιτούν άμεσες και ταχείες παρεμβάσεις. Η νομοθεσία βεβαίω σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι ενδιάμεσοι, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε ώστε να κάνουμε στοχευμένες δράσεις. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω εδώ και να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν Περέιρα ή ο άλλος συνάδελφος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Πασχόλησης για Διεθνείς Υποθέσεις και ο συνάδελφος ε, θα πάρει το λόγο στη συνέχεια γιατί έχουμε και μια σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση για τους εργαζομένους από τη Βόρεια Κορέα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Το γνωρίζουμε. Η Κομισιόν ε, είναι σε επαφή με πολλά κρατημέλη για το θέμα αυτό. Όμως, έχω και μια ερώτηση για τον ε, καθηγητή Μπρούκερ γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό το καθεστώς των κυρώσεων πρόσφατα εξέδωσε μία απαγόρευση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν άδειες εργασίας σε βορειοκορεάτες. Υπάρχει απόλυτη απαγόρευση λοιπόν. Η ερώτησή μου είναι δεν γίνεται σεβαστή η απαγόρευση αυτή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και έχω άλλες δύο παρατηρήσεις ε, για τους ε, οικιακούς εργαζομένους και για την ε, οδηγία εμπορίας ανθρώπων. Για τους οικιακούς εργαζομένους, η Κομισιόν έχει συστήσει τα κράτη-μέλη να κυρώσουν την Σύμβαση Εργασίας του ΔΟΕ κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Υποστηρίξαμε τη ΔΟΕ και θέλουμε ουσιαστικά να επικυρωθεί ε, η σύμβαση αυτή. Επίσης έχουμε συστήσει και στα κράτη-μέλη να την επικυρώσουν, θα επικυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε οργανώσει συναντήσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για να δούμε αν μπορούν να υπάρχουν κάποια εμπόδια για την επικύρωση. Επίσης οργανώνουμε και μια συνεδρίαση με το ΔΟΕ και τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ε, επαγγελματική ε, ασφάλεια με την επικοινωνική ασφάλεια και την υγεία. Επίσης, ε, εμείς ε, έχουμε υποστηρίξει τη δουλειά της ε, για, την, για ένα νέο πρωτόκολλο και όταν υιοθετήθηκε αυτό, με την υποστήριξη της Ένωσης, ζητήσαμε τα τη μελη να επικυρώσουν το πρωτόκολλο το συντομότερο και πάνω από τα μισά κράτη-μέλη έχουν ήδη κυρώσει το πρωτόκολλο και τα υπόλοιπα προετοιμάζουν την κύρωση. Είναι ένα σημαντικό πρωτόκολλο αυτό και ελπίζουμε ότι θα σημαίνει και μία διαφορά στην πράξη στα νομικά συστήματα. Συνάδει πάρα πολύ με την οδηγία της Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων. Είναι ένα σημαντικό έγγραφο, το οποίο έχει υποστηρίξει το έργο της ΔΟΕ στον τομέα αυτό. Δύο παρατηρήσεις ήταν αυτές, αλλά έχω και μια ερώτηση, όπως είπα, στον καθηγητή Μπρούκερ για τους ε, εργαζομένους από τη Βόρεια Κορέα. Και κατόπιν, ο συνάδελφος ο Φερνάντο Βάσκες ε, θα πάρει το λόγο για την ιστορική διάσταση. Καλείτε τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω ότι η εκμετάλλευση στην εργασία υπάρχει σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους. Επίσης, ε, να σας πω ότι υπάρχει και σε καθαρά εθνικές ε, περιπτώσεις εγώ. Ως ε, αρμόδιος για την απόσπαση των εργαζομένων, γνωρίζω ότι όταν υπάρχει ένα διασυνοριακό στοιχείο, αυτό κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση. Η έλεγχη είναι πιο πολύπλοκη. Όμως είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιήσουμε ότι δεν αποτελεί αυτό την πηγή του προβλήματος. Απλώς καθίσταται πιο πολύπλοκο το πρόβλημα. Ο έλεγχος ουσιαστικά είναι αρμοδιότητα εθνική και όταν υπάρχει ένα διασυνοριακό στοιχείο γίνεται στη χώρα υποδοχής όπου λαμβάνει η χώρα η εργασία όμως ε, πολλά στοιχεία είναι απαραίτητα Πολλέ πληροφορίε είναι απαραίτητε που δεν μπορούν να βρεθούν παρά ίσω ε, στη χώρα προέλευση του εργαζομένου. Για του επιθεωρητέ ε, λοιπόν ε, εργασία, όταν μιλάμε για αποσπασμένου εργαζομένου, η πρόκληση είναι η συνεργασία με τι αρμόδιε εθνικέ αρχέ του κράτου μέλου προέλευση. Αυτό κάνει πιο πολύπλοκα τα πράγματα, όμως θέλαμε να είναι δυνατόν μέσω μιας οδηγίας του 2014 η οδηγία εκτέλεσης ε, στο θέμα της απόσπασης ε, που θέτει κάποιες υποχρεώσεις για την επιθεώρηση αλλά προβλέπει και μια σειρά διοικητικών μέτρων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με μια σειρά προθεσμιών που πρέπει να γίνουν σεβαστές ε, προκειμένου να δοθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθεται από το κράτος μέλος υποδοχής. Αυτό δεν θα λύσει βέβαια όλα τα προβλήματα αλλά κυρίως στον τομέα της απόσπασης είναι σημαντικό να φτάσουμε στην ε, κατάσταση όπου οι εθνικές ε, διοικήσεις των δύο κρατών επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. κυρία Μωράν Σαρτιέ ανέφερε την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Είναι μια πρόταση που έχει υποβάλει η Κομισιόν και σκοπεύει ακριβώς στο να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικήσεων, να θεσπίσει κοινά συστήματα επιθεώρησης και σίγουρα θα αποτελεί σημαντική συνεισφορά στον τομέα. Θα αναφέρω επίσης την πλατφόρμα για την δηλωμένη εργασία, γιατί συχνά έχουμε αναφέρει τους, την αδήλωτη εργασία, συγγνώμη, γιατί συχνά αναφέρουμε του αποσπασμένου εργαζομένου, αλλά έχουμε και το θέμα τη αδήλωτη εργασία. Η πλατφόρμα ήδη έχει παρουσιάσει αρκετά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχει φέρει σε επικοινωνία τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, μπορούν να ανταλλάξουν γνώσεις και επίσης υπάρχουν και πολλές μανέτες που ανέφερε και η κυρία Μωράν Σαρτιέ που έχουν ε, ήδη γίνει αλλά θα γίνουν και στο μέλλον. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό να αναφέρουμε και αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο για να δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Θα έλεγα τώρα να δώσουμε το λόγο με την ανάποδη σειρά. Να δώσουμε δύο-τρία λεπτά στον καθένα για να μπορείτε να απαντήσετε. και ίσω και να εξαγάγετε και κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τόσο υπόθηκαν από την Κομισιόν. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ιουλιάνο. Μάλιστα. Εγώ τελείωσα να ξεκινήσω. Να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρέμβασή τη. Μα έδωσε μια σειρά ξεκάθαρων στοιχείων σε σχέση με τις δεσμεύσεις και τις Κομισιόν απέναντι στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας Η κυρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έφυγε τώρα μίλησε για το ότι πρέπει να αναγνωριστούν περισσότερο οι συλλογικές συμβάσεις ως ένα από τα μέσα αναχέτησης, αντιμετώπισης κάποιων φαινομένων που σχετίζονται και με την καταναγκαστική εργασία. Και φυσικά όλη η δουλειά που γίνει σε κάποιες χώρες ε, λόγω της μαύρης ε, εργασίας ε, να ξεπεραστούν οι επισφαλείς καταστάσεις εργασίας. Σήμερα έχουμε κάποιες μορφές, επικίνδυνες μορφές μάλιστα εκμετάλλευσης. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο λοιπόν θα ήταν ένα κεντρικό στοιχείο. Επίσης ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που μας ανέφερε το σημαντική συνάντηση που έχουμε. Θα είναι η εκατοστή επέτειο της ίδρυσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και φυσικά θα δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα σημαντικό ραντεβού γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των νομοθετημάτων της αλλά και της ικανότητάς της ε, να απευθύνεται σε 27-28 κράτη-μέλη σε σχέση με την επικύρωση αυτών των συμβάσεων ε, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη και αν ε, θα έχουμε τις εκλογές, Ίσως θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη νέα θητεία υπό το φως ενός πολύ σημαντικού και κεντρικού ζητήματος. Και το περιλαμβάνω για να μπορέσει να επιβιώσει και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντίρινγκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πολύ ξεκάθαρα το εξή. Ο Μπεν Ράσελ είπε ότι τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου δεν είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με το τι ξέρουμε, αλλά με το τι κάνουμε. Και περί αυτού πρόκειται. 800 συνεντεύξει έκανα σε πάνω από 30 ε, ομάδε κτλ. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε αρκετέ γνώσει, έχουμε μια σαφή εικόνα τη κατάσταση, αρκετά ακριβή εικόνα σε ό,τι αφορά τη γεωργία, ε, τι γίνεται στους αμπελώνες, ε, στις οικοδομές, ε, στους δρόμους λοιπά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε τώρα είναι γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και εμένα με κάλεσαν σε μια παρουσίαση PowerPoint επικεφαλής της Ευρωπαϊκής στην Αυστρία και μου έδειξαν πολύ ωραίες εικόνες αξιοθρύνητων συνθήκων εργασίας για κάποιους εργαζόμενους και μου ε, είπε ότι κανένας δεν αναφέρει αυτές ε, τις περιπτώσεις στην αστυνομία επειδή φοβούνται. Οι άνθρωποι πληρώνουν τις εισφορές τους, αλλά δεν ε, γίνονται σε αυτά τα δικαιώματά τους. Υπήρξαν επιθεωρητές που μας είπαν ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο χώρος εργασίας. Αν είναι αυτός υγιής και ασφαλής, όχι οι εργαζόμενοι. Επίσης, κάποιοι μου είπαν θα θέλαμε να συλλέξουμε στοιχεία, αλλά πώς, δεν ξέρουμε να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία. δεν ξέρουν πώς να συλλέξουν πληροφορίε που θα μπορούσαν να τις δώσουν στις αγγελικές και αστυνομικές αρχές στη συνέχεια. Επομένω υπάρχουν πολλά ε, κενά και εκεί δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο, γιατί δεν υπάρχουν ε, δίκες σχετικές, ε, γιατί δεν προσφέρουν στα δικαστήρια. Μα γιατί δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη τα θύματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και εκεί μπορεί να ξεκινήσει η δράση μας, αλλά μπορεί να ξεκινήσει ε, και σε άλλα επίπεδα, δημόσιες προμήθειες για παράδειγμα. Είχαμε στην Ελλάδα μία περίπτωση ε, με σοβαρή εκμετάλλευση από μία εταιρεία ε, κατασκευαστική οδικά έργα. Συγκεκριμένα ήταν το αντικείμενο και παρότι αποδείχθηκε ότι υπήρχε σοβαρή εκμετάλλευση. Η σύμβαση δεν έλεγε τίποτα για τις συνθήκες εργασίας, άρα δεν μπορούσαν ε, να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι πολλά ε, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει με το λεγόμενο social branding, αλλά αυτό δεν υπάρχει ακόμη. Fair trade υπάρχει, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τις ε, μάλλον έχει να κάνει και με τις συνθήκες εργασίας, αλλά πρέπει να υπάρξει και ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Ο κόσμος να ξέρει τι αγοράζει. Δεν θα αγόραζε ρούχα που έχουν φτιάξει παιδιά τα οποία είναι αντικείμενα εκμετάλλευση ε, ε, και δουλεύουν υπό απαράδεκτες συνθήκες. Αυτά θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο, η κυρία Τέκουη. Συμφωνώ απόλυτα. όσα υπόθηκαν πριν από κάποια χρόνια αποκτήσαμε την επαρκή νομοθεσία έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Όμως ένα από τα παραδείγματα που μπορώ να σας αναφέρω στην Ισπανία, το χάρη, έχουμε τις εργαζόμενες ε, για τη συλλογή της ε, φράουλα. 50.000 ε, άτομα έρχονται από το Μαρόκο και από άλλες χώρες Ευρώπης να κάνουν αυτές τις δουλειές. Υπήρχε ένα άρθρο από το γερμανικό τύπο ότι υπήρχαν βιασμοί και σεξουαλική παρενόχληση και όλα αυτά ουσιαστικά δημιούργησαν ένα τεράστιο κίνημα έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι συνεχίζουν να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, ναι έχουν ε, σημειωθεί ε, ουσιαστικά πολύ μεγάλες βελτιώσεις, όμως ε, συνεχίζουμε να έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Γιατί ουσιαστικά τα άτομα αυτά δεν προφέρουν σε καταγγελίες γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους για την επόμενη εποχή συλλογής της φράουλας γιατί όταν ε, ε, ουσιαστικά κάνουν την καταγγελία ήδη έχουν επιστρέψει στη χώρα τους. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα γιατί όλα τα θέματα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών, την ε, σεξουαλική παρενόχληση κτλ. είναι πάρα πολύ λεπτά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεικτούν. Κάποια συνδικάτα που κατήγγυλαν την κατάσταση ε, ουσιαστικά δέχτηκαν και αυτά καταγγελίες με τη σειρά τους από τους ε, ε, εργοδότες. Θέλω να απαντήσω στο Χαβιέρ για τις ερωτήσεις που έθεσε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Όλοι βρισκόμαστε πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα το εξής. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει ο κόσμος της εργασίας με τέτοιο τρόπο που τα εργαλεία που έχουμε μέχρι τώρα δεν μας ε, φτάνουν πια. Σε ποιες ε, πτυχές. Το πρώτο είναι στο να δούμε τι σημαίνει εργαζόμενος. Αυτό ε, ουσιαστικά έχει διαραγεί. Δηλαδή, ε, όλο ένα και πιο ευρύνεται τα σύνορα για το τι σημαίνει μισθωτός. Επίσης πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει επιχείρηση. Δεν μπορούμε ε, ουσιαστικά να καλύψουμε ε, τις ε, δυσκολίες και την πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Θα πρέπει να εργαστούμε και για το πώς θα κάνουμε μια ρύθμιση σε σχέση με τους μισθούς. Θα πρέπει να εργαστούμε σε μια παραλληλόδο που έχει να κάνει και με τον ελάχιστο μισθό, με τον κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι είναι κάτι απαραίτητο. Και φυσικά είναι πολλή δουλειά ακόμη και σε αυτό το τομέα που πρέπει να γίνει. Έχουμε και το ελάχιστο εισόδημα. Νομίζω ότι αυτό βρίσκεται στην πολιτική ατζέντα σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και λυπάμαι πολύ που δεν είναι εδώ η βουλευτής που έκανε την ερώτηση για τις γυναίκες. Γιατί θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Αυτή αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι ε, ουσιαστικά να αναγνωριστούν στην αγορά εργασίας ε, τα πτυχία ε, των ε, νέων. Επειδή έχουμε εντελώς διαφορετικές επιλογές ακόμη και το 2018 από τους νέους και τις νέες και πρέπει να δούμε τι ακριβώς σπουδάζουν, ποια ειδικότητα διαλέγουν για να δούμε ότι είμαστε υπερβολικά μπλεγμένοι ακόμη κολλημένοι στα στερεότυπα και στα κλισέ. Εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη πλαισίωση, επομένως χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις για τον εκπαιδευτικό και εργασιακό προσανατολισμό, έτσι ώστε οι νέες τα παιδιά να μπορούν να ανοίξουν τις δυνατότητές τους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό γιατί φυσικά όλο αυτό καθορίζει και την αγορά εργασία και ευνοεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και κάτι τελευταίο. Ιδίω έχοντα κατά νου ότι αν καταλάβουμε, ένουμε, αν θεωρούμε ότι ο κόσμος θα γίνει όλο ένα και πιο παγκοσμιοποιημένος και η ψηφιοποίηση θα έχει πολύ σημαντικό βάρος, οι δυσκολίες που έχουν τα κορίτσια για την πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα θα πρέπει να μας ανησυχούν πάρα πολύ γιατί αν δεν καταφέρουμε να υπάρχει μία πιο άμεση πρόσβαση των κοριτσιών στην τεχνολογία, στο μέλλον θα βρεθούμε στο να έχουμε ένα νέο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, Ευχαριστώ. Ο καθηγητής Μπρέουκερ. Thank σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνοντας θα απαντήσω στο ερώτημα της Επιτροπής που ήταν απλό. Δεν έχω όμως σας δώσω μια απλή απάντηση. Υπάρχει οδηγία που δεν επιτρέπει την πρόσληψη βορειοκορεατών πλέον Έχουμε δει αυξητικέ αλλαγέ, έχουν γίνει διάφορα, εκθετικέ αλλαγέ μάλλον, έχουν γίνει διάφορα έκτοτε. Το 17 είδαμε κάποια ζητήματα. Και με βάση τις κυρώσεις υπάρχει μια περίοδος χάριτος μέχρι το 19. Οπότε και θα πρέπει να έχουν φύγει όλοι οι Βορειοκορεάτε εργαζόμενοι και οι κοινοπραξίες. Θα πρέπει να έχουν διαλυθεί ήδη πιο πριν. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, εξ όσων γνωρίζω. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα έλλειψη δεδομένων όμω. Για τρία χρόνια έχω κάνει έρευνα. Είμαι πολύ ενό κράτου μέλου τη Ένωση. Παρ' όλα αυτά, δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να συγκεντρώσω τα στοιχεία τα οποία υποτίθεται θα μπορούσα ε, να προσποριστώ. Γιατί είναι δημόσια δεδομένα, στα οποία θα έπρεπε να έχω πρόσβαση κανονικά. Και μήνυση Μάλλον αν κάνω μήνυση μόνο έτσι θα μπορούσα ίσως ε, κάποια αγωγή. Για τη χώρα μου, την Ολλανδία, είναι πιο δύσκολα. Ε, και ακόμα και από την Πολωνία που έχει καλύτερη πολιτική. Ίσως δούμε και κάποια ελάφρυση των ποινών, των προστήμων σε τέτοια Βορεια Οπότε κάποιοι ίσω να μπορούν να ξαναέρθουν να εργαστούν από τη Βορεια Κορέα στην Ευρώπη. Και έτσι θα ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Που θα είναι και πάλι στο έλεος των εργοδοτών τους αυτοί οι εργαζόμενοι. Στηρίζω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι δύο μιλητέ. Απλά υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά του Βορειοκορεάτε. Εκεί ε, Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν είναι τόσο ασαφή και θολά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό που θα έπρεπε να έχουν με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. κτλ. Άρα είναι θέμα εφαρμογής της νομοθεσίας. Δεν είναι βέβαια τόσο απλά στα, τα πράγματα στην πράξη. Αλλά από ό,τι έχω δει, παραδείγματο χάρη εκτό θεωρήσεων διαβατηρίου για εργαζόμενου από τη Βόρεια Κόρεα, αυτό έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται ακόμη και αφού η κυβέρνηση ότι θα πάψει να ε, εκδίδει θεωρήσει. Αλλά δεν το έχει κάνει, αν δείτε τα στατιστικά. Συνεχίζει και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μόνο η λόγο κυβέρνηση θα μπορούσε να το απαντήσει. Αυτά λένε τα στατιστικά μας όμως. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αντιβαίνει στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι δικηγόρος. Δεν είμαι νομικός. Δεν μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν. Παρά την προσοχή όμως από τα μέσα ενημέρωσης και τα ε, ερωτήματα που θέτετε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκμετάλλευση των Βόρειο-Κορεατών στην Πολωνία και άλλες χώρες συνεχίζεται. Στου τελευταίου μήνε βέβαια δεν έχω ελέγξει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει η κατάσταση ε, αλλάξει από τότε που σταμάτησε το project αυτό πριν από κάποιου μήνε. Bene. Ωραία. Τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες που μας βοήθησαν να προσεγγίσουμε πιο συγκεκριμένα αυτό το θέμα. Τελειώνει εδώ η συνεδρίασή μας. Επόμενη συνάντηση στις 28 του Ιούνιου από τις 9 μέχρι τις 12.30 εδώ στις Βρυξέλλες. Καλό βράδυ και γεια σας.